Από την ανάγκη θεωρήσεως των διαβατηρίων των πολιτών του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Δίας Ντεμέρα για τρία λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε μερικοί από εσάς, Ήμουν ε, εισηγητής του κανονισμού 539-2001 που ρυθμίζει την πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν επίσης ε, για το μηχανισμό αναστολής που απορρέει από τον ε, κανονισμό αναφοράς. Και επανειλημμένως συμμετείχα στη συμπερίληψη των αρνητικό κατάλογο του κανονισμού διαφόρων χωρών όπως η Κολοβία, το Περού, Ταϊβάν, Γεωργία, Ουκρανία κτλ. Όλες αυτές οι χώρες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι κυρίαρχες χώρες, είναι κυρίαρχα κράτη. Η πρώτη φράση στο άρθρο 1, εδάφιο 1 του κανονισμού 539 αρχίζει ως εξής. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών κτλ. κτλ. Στην ε, συζήτηση που έχουμε σήμερα δεν μιλούμε για καμία χώρα. Για μας το Κωσυφοπαίδιο είναι σερβική επαρχία, όπως η Βοηβοδίνη και ανήκει στην σερβική κρατική επικράτεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να διευκολύνουμε πολιτικά εργαλεία που διευκολύνουν τη διαμέληση ενός κυρίαρχου κράτους όπως είναι η Σερβία. Και η θέση μας ως Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα είναι γνωστή της Πάσης η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζεται από 28 χώρε. Ο κανονισμό ισχύει για 28 χώρε, όχι για 23 χώρε. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν να εφαρμοστεί εν μέρη ο κανονισμό. Θα ήταν πολύ αμφίβολη νομιμότητα σε ένα τέτοιο μέσο νομικό. Και η νομοθετική πρωτοβουλία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Σλοβακία, ούτε στην Κύπρο, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στην Ελλάδα. Γιατί αν ευοδοθεί αυτή η πρόταση, σίγουρα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δεχθεί αγωγές και στάσεις από τις πέντε ε, κυρίαρχες χώρες που προανέφερα. Γιατί καμία από αυτές τις πέντε χώρες δεν θα επιτρέψει την ε, απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης των κατοίκων μιας σερβικής επαρχίας. Δεν δίνουμε θεωρήσεις σε κατοίκους μιας επαρχίας, μόνο σε υπηκόους κυρίαρχων χωρών. Και αυτό που λέω είναι και νομικός και δικαστικός, αναφυσβήτητο και αδιαφιλονίκητο και πολύ λιγότερο από τον κανονισμό 539 κάθετος του 2001. Τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις με μπλε κάρτα έχουν υποβληθεί από την κυρία Βερζία και από την κυρία Φαγιόν. Τις δέχεστε κύριε Διαζεμέρα. Μάλιστα, πρώτα η κυρία Βερζιά και μετά η κυρία Φαγιόν. Παρακαλώ, κυρία Βερζιά. Κύριε Ντίας Δεμέρα, γνωριζόμαστε, συχνά συνεργαζόμαστε και ξέρω ότι είστε εξαιρετικό νομικός. Γνωρίζετε ότι οι πέντε χώρες που αναφέρατε έδωσαν την, το OK για την απελευθέρωση των θεωρήσεων άσχετα με το θέμα της αναγνώρισης του κωσυφοπεδίου. Ε, οπότε τι γίνεται με τον ΟΗΕ και την αναγνώριση των ε, χωρών και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών. Δεν δίνεται καμία αξία σε όλα αυτά. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Βεργζία. Και εγώ έχω εξαιρετική γνώμη για σας και το έργο σας. Αλλά φαίνεται δεν είστε καλά πληροφορημένοι. Οι πέντε χώρε μέλη δεν έδωσαν ε, την έγκρισή του σε κάτι που δεν δύναται να δώσουν την έγκρισή του. Οι πέντε χώρε μέλη δεν μπορούν εν μέρη να χορηγήσουν απαλλαγή αποθεωρήσει σε μια επαρχία που ανήκει σε μια κυρίαρχη χώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαγιό έχει να θέσει ερώτηση με μπλε κάρτα. Αγαπητέ Αγκουστίν, και εγώ έχω εξαιρετική συνεργασία μαζί σου και γνωρίζω ότι είσαι νομομαθής και επαΐων στα νομικά ζητήματα. Αλλά και εγώ είχα επαφή και με εκπροσώπους και των πέντε χωρών που δεν αναγνώρισαν το κοσυφοπαίδιο και μάλιστα δίκαιο έχει συνάδελφος. Αναγνωρίζουμε ταξιδιωτικά έγγραφα και όχι υπηκότητα. Οπότε δεν είναι ε, θέμα ε, μπορεί κάποιο να συμφωνήσει με την απελευθέρωση χωρί να έχει αναγνωρίσει το κοσυφοπέδιο. Άλλωστε, το 2009 συμφωνήσαμε να απαλλάξουμε του υπηκόου τη Ταϊβάν από την υποχρέωση θεώρηση. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναγνωρίσει το κράτο τη Ταϊβάν, την Ταϊβάν ω κράτο, ω ανεξάρτητη χώρα. Κυρία Φαγιό. Και εγώ αναγνωρίζω και εκτιμώ ιδιαίτερο το έργο σας και τη συνεργασία που έχουμε κατά καιρούς. Η απάντηση που θα σας δώσω είναι παρόμοια με αυτή που έδωσα προηγουμένως στην κυρία Βερζιά. Άλλο είναι η διευκόλυνση ενός ταξιδιωτικού εγγράφου και άλλο πράγμα είναι η χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου σε κάποιον που στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων δεν είναι υπήκος κυρίαρχης χώρας. Επαναλαμβάνω και διατρανώνω ότι από νομική άποψη και άσχετα αν την έχουν αναγνωρίσει πολλές χώρες από την ε, διεθνή κοινότητα, ο συγκεκριμένος κανονισμός ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για τις 23 μόνο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε από νομική άποψη δεν μπορεί να εφαρμοστεί με, μερικός μόνο, εν μέρη μόνο ο κανονισμός. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα ασκηθούν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τις 5 χώρες που δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό και δεν δεσμεύονται γιατί δεν αναγνωρίζουν τη σερβική επαρχία που συνιστά το κοσυφοπαίδιο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μάμικινς για 1,5 λεπτό. Αντρέης, έχετε το λόγο. Επίτροπε, αξιότιμα μέλη, το κοσυφοπαίδιο αποκλείστηκε από το καθεστώς ε, την προηγούμενη δεκαετία, ενώ άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είχαν αυτό το προνόμιο. Μπορεί να ερμηνεύουμε την ιστορία της χώρας ε, διαφορετικά, αλλά δεν μπορεί να είναι πολιτική, πολιτικ, η χώρα αυτή. Η, το Κωσυφοπαίδιο χρειαζόταν την ε, διαδικασία, το καθεστώς απαλλαγής μετά την ε, διακήρυξη της Θεσσαλονίκης. Εμείς περιμέναμε μέχρι ότου το Κωσυφοπαίδιο εκπληρώσει 95 ε, σημεία αξιολόγηση και το έκανε. Ε, πώς λοιπόν μπορούμε τώρα να στερήσουμε το δικαίωμα που έχουν. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι δίκαιη, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ε, υποσχέσεις. Το 95% των Κωσοβάρων είναι υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αυτό θεωρήσουμε ως μελλοντικό κράτος μέλος. Δεν είναι δυνατόν να υπονομεύομαι, υπονομεύομαι το μέλλον μιας φιλοευρωπαϊκής χώρας και ε, εύχομαι ε, να ε, εκλείψει αυτή η άδικη μεταχείριση της χώρας αυτής. Επίσης, ε, το, η ε, Δύση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό από το Κωσυφοπαίδιο. γι' αυτό στηρίζω την εισηγήτρια κυρία Φαγιών και σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο, η κυρία, κυρία Τόμας έχει το λόγο, εκ μέρους τη ΣΥΑΡ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς, προς τους υπηκόους τρίτων χωρών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη χώρα αυτή στενό εταίρο το να μιλούμε για την ευρωπαϊκή προοπτική του Κωσυφοπεδίου και ταυτόχρονα επιμένουμε για θεωρήσεις για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη υποκρισία. Πολλό δε μάλλον είναι υποκρισία να υποκινείται από πολιτικά κίνητρα, ενώ ακούμε την ιστορία για τα κριτήρια που είναι σημαντικό να εκπληρωθούν. Αν είναι σημαντικά τα κριτήρια, που εγώ θεωρώ ότι είναι, τότε θα πρέπει στην περίπτωση που η χώρα πληρεί τα κριτήρια να μην υπάρχουν πια εμπόδια. Μια όμως και πρόκειται για το κοσυφοπαίδιο, υπάρχει πάλι πρόβλημα με το διεθνέ καθεστώ τη χώρα αυτή. Έχουμε κάποιε χώρε μέλη που ακόμη δεν έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο. Είτε μα αρέσει όμω είτε όχι, το Κωσυφοπαίδιο είναι μια χώρα. Στο χέρι μα είναι να τη βοηθήσουμε να γίνει σταθερή και ευημερούσα χώρα, συντροφική και φιλική, και αντί να τη σαμποτάρουμε από εγωισμό, υποκρισία και πολιτικαντισμό. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Τόμασιτ. Μία μπλε κάρτα. Ε, από τον κύριο Ρούμπιχ έχει υποβληθεί. Τη δέχεστε? Αγαπητοί συνάδελφε, υπάρχει μια ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε από τον κύριο Ρούμπιχ. Τη δέχεστε? Μπείτε σεν, κύριε Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό να δούμε τα κριτήρια που έχουν εκπληρωθεί. Όντως, τι σχέση έχει αυτό με την ε, ε, άδεια παραμονής. Αυτά τα δύο τα διαφοροποιούμε. Η θεώρηση είναι πολύ σημαντική για να, ε, να διευκολύνουμε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάδελφε, πιστεύω ότι εδώ πρόκειται για πολιτικατισμό. Χώρες με πολύ περισσότερους εγκληματίες, με πολύ χειρότερη κατάσταση διαφθοράς, ε, τους ανοίξαμε τις ε, πύλες και καταργήσαμε τις θεωρήσεις. Ενώ στο Κωσυφοπέδι δεν το κάναμε. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί πολιτικαντισμό, καθαρό πολιτικαντισμό. Ευχαριστώ. Το λόγο κύριο Σελίμοβιτς τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω από τη συζήτηση αυτή. Συχνά επικρίνουμε χώρες γιατί δεν ανταποκρίνονται στις ε, προϋποθέσεις. Κάνουν, λένε το ένα, κάνουν το άλλο. Ε, εν εμείς φερόμαστε όπως οι χώρες αυτές. Πώς είναι δυνατόν αυτό. Έχουμε θέσει συγκεκριμένες απαιτήσει για να εκπληρώσει το κοσυφοπαίδιο. Ε, οι απαιτήσει ε, ε, υπαγορεύτηκαν από όλε τι χώρε και αυτέ που δεν αναγνωρίζουν το κοσυφοπαίδιο. Και το κοσυφοπαίδιο το αποκρίθηκε. Η Κομισιόν έκανε την αξιολόγηση, είπε ότι ναι, εκπληρώθηκαν οι προποθέσει. Και τώρα η απάντησή μα είναι Τίποτα. Νομίζω ότι αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία μας. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε ή ε, να βάλουμε και άλλες προϋποθέσεις. Δεν το κάναμε. Όμως όλες οι προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί. Γι' αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να σταματήσει ε, την κοροϊδία και να προχωρήσει στην απαλλαγή γιατί αυτό πράγματι ε, υποσκάπτει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπίλντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ κυρία το να ράψουμε ένα ανοιχτό, μια ανοιχτή πληγή με το αίτημα για την απελευθέρωση των θεωρήσεων ότι, φαίνεται ότι κάνουμε κατάχρηση της υπερβολής. Το να ζητούμε όμως μια αξιοκρατική απόφαση, ενώ το τελευταίο καιρό η κοσυφοπαίδεια φαίνεται, το κοσυφοπέδιο φαίνεται ότι παίζει με τη φωτιά. Τι να πούμε για, τις, ε, για τους δασμούς 100% από τις σερβικές εισαγωγές εις βάρος της ε, ε, Κεντροευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ή η μετατροπη των δυνάμεων ασφαλείας σε στρατό στο κοσυφοπέδιο κατά παράβαση των θεμελιωδών κειμένων. Και ενώ χύνουμε δάκρυα για την απομόνωση του ε, τι γίνεται με, τη, με την σερβική μειονότητα και την καταπάτηση των υποχρεώσεων για τους σερβικούς δήμους που έχουν μείνει κενό γράμμα παρά τη συμφωνία του 2013. Το Κωσυφοπέδη όλο και απομακρύνεται από την ενταξιακή του πορεία και επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να είναι ένα άναρχο κράτος στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Επίρου. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μάντλ για δύο λεπτά. Παρακαλώ κύριε Μάντλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι ε, μιλώντας υπέρ τη απελευθέρωσης των θεωρήσεων για το κοσυφοπαίδιο, κατ' ουσίαν μιλάω εξ ονόματο της πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, γιατί έχουμε ήδη ψηφίσει υπέρ τη απελευθέρωσης και τώρα εναπόκειται στο ε, Συμβούλιο να εκπληρώσει μια υπόσχεση της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ε, τα κριτήρια καλύφθηκαν από το κοσυφοπαίδιο. Όλοι μα γνωρίζουμε ότι είναι έξι κράτη στην νοτιοανατολική Ευρώπη και ε, μόνο το 10% των 80 εκατομμυρίων, το 1,8% δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει ελεύθερα. Οι ε, κάτοικοι του Κοσμοπεδίου θα πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα και παρεπιπτόντως όλοι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την διαφθορά, να έρθει το κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα, να βοηθήσουμε τους πολίτες της χώρας αυτής να μπορούν να βρουν δουλειά, εκπαιδευτούν στην πατρίδα τους. Το θέμα δεν είναι να φεύγουν για να ψάχνουν να βρουν αλλού δουλειά στην Ευρώπη. Αυτό που έχει σημασία είναι να ταξιδεύουν ε, χωρίς ε, ε, τις θεωρήσεις, χωρίς χρονοκαθεστερήσεις. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό για τις οικογένειες. Αυτό σημαίνει απελευθέρωση των θεωρήσεων και πιστεύω ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζει τους πολίτες του Κοσφοπεδίου, στους οποίους αξίζει η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάντλ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πίκουλα για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ κύριε Πίκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων του κοσυφοπεδίου έπρεπε να είχε ήδη ε, λάβει χώρα. Γιατί έχουμε, τέσσερα χρόνια μετά τις υπόλοιπε χώρε των Δυτικών Αλβανίων. 95 κριτήρια χρειάστηκε να εκπληρώσει το Κωσυφοπέδιο μέχρι το 2016 και δύο επιπλέον κριτήρια για το κράτος δικαίου και την πάταξη της διαφθοράς. Τα πιο δύσκολα όπως η ε, κύρωση πριν από ένα χρόνο της συνοριογραμμής με το Βούνιο. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν έγινε από τη δικιά μας πλευρά. Εξακολουθούμε να απομονώνουμε τα, τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου που είναι η χώρα με τον πιο νεαρό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να μας ευνηδιάζουν οι δασμοί που επέβαλε το Κωσυφοπέδιο ε, στα εισαγόμενα προϊόντα από τη Σερβία και τη Βοσνία θα πρέπει όλα αυτά να τα εκλάβουμε στο πλαίσιο της δυσαρέσκειας του κοσυφοπεδίου με μια παράδεκτη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ε, συνεπής και να σέβεται τις αρχές που ήδη επέβαλε. Θα πρέπει να μην πολιτικοποιούμε αυτό το θέμα και να το συνδυάσουμε με τις νόμιμες και προταξιακές διαδικασίες. Θα πρέπει επιτέλους να γίνουν οι κάτοικοι του Κωσυφοπεδίου ισότιμοι με τους υπηκόους των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί πραγματικά το αξίζουμε τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο και ο κύριος Κολομπιέ. Κύριε Πρόεδρε, ακόμη και σήμερα πέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δικαίω αρνούνται να αναγνωρίσουν το κοσυφοπαίδιο ω ε, ανεξάρτητο κράτο. Η ανεξαρτησία άλλωστε του κοσυφοπαιδίου δεν είναι παρά η απόρρεια των βάρβαρων βομβαρδισμών του σερβικού λαού πριν από 20 χρόνια και του επεμπλουτισμένου ουρανίου που υπάρχει. Η απαλλαγή από τις θεωρήσεις για τους κατοίκους του Κωσυφοπεδίου θα ήταν ένα επιπλέον βήμα ε, στην ανταξιακή του πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που απορρίπτουμε επισήμως πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τα κριτήρια. Εγώ βλέπω ένα κριτήριο, την απαράδεκτη μεταχείριση ή την απαράδεκτη συμπεριφορά της κοσοβάρικης κυβέρνησης προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, έχουμε ένα ψευδοκράτος, ε, μαφιόζικο και εξισλαμισμένο, που όπως λέει το, μια έκθεση του State Department, ε, ε, προβαίνει σε θεσμικέ μεταρρυθμίσει ε, για την απασχόληση και τι κοινωνικέ υπηρεσίε, ε, προβαίνει σε εκφοβισμού και επιθέσει και θέλει να απαγορεύσει τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου να ασκήσουν τη θρησκευτική του ελευθερία. Οπότε θα ήθελα να πω στην εισηγήτρια της έκθεσης ότι το εγχείρημά της δεν είναι σωστό. δεν πρόκειται να βοηθήσει την επανασυμφιλίωση των λαών της πρώην Ιουκοσλαβία που είναι της πρώην που είναι όλοι λαοί, φίλοι λαοί. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, συνάδελφοι. Να σέβεστε όμως το χρόνο, γιατί 25 δευτερόλεπτα παραπάνω είναι πολλά. Δεν θέλω να σας διακόπτω, αλλά θα με αναγκάσετε να το κάνω. Το λόγο έχει η κυρία Γουόρτ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, κυρία Γουόρτ. Έχει φτάσει η στιγμή έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να τηρήσουν την υποχρέωσή τους, να επιτρέψουν στους Κωσοβάρους να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεώρηση. Το Κωσυφοπαίδιο είναι μια νέα χώρα που έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες μετά από τις ε, ιδεχθείς ε, εθνοκαθάρσεις ε, προσπάθησε το Κωσυφοπαίδιο να προσαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσει την απελευθέρωση και θέλω να πω ότι και οι προϋποθέσεις δεν ήταν ίδιες για όλους. Άλλοι ε, μπόρεσαν να τα πετύχουν ε, γρηγορότερα. Εγώ αυτό το βρίσκω άδικο για τους Κωσοβάρους. Ε, ε, με τακτικές επαφές με την κοινωνία των πολιτών, κυρίως με τους νέους και τις γυναίκες. Με αυτή την ευκαιρία είδα πολίτες που επιθυμούν διακαώς να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μπλοκάροντας τη διαδικασία απελευθέρωση των θεωρήσεων, το Συμβούλιο στέλνει λάθος μήνυμα. Πολλοί νέοι κοσοβάροι είναι απογοητευμένοι και αισθάνονται ότι τους έχει εγκαταλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήλπιζαν να ενταχθούν σε αυτό το ευρωπαϊκό ειρηνικό εγχείρημα, αλλά σιγά σιγά η ελπίδα τους εγκαταλείψει Πού θα στραφούν λοιπόν, φοβάμαι και θα ήθελα να πω κάποια ε, που άκουσα σήμερα το βράδυ με φόβησαν. Εγώ ως ε, Βρετανίδα ε, βουλευτής, ευρωβουλευτής, έχω κοσοβάρους στο δικό μου, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, στο Μάντσεστερ. Αυτή είναι πρόσφυγες πολέμου συμβάλλουν στην κοινωνία μας και αν τους εγκαταλείψουμε εγκαταλείπουμε όλους κοδοπάρους και αν το κάνουμε ντροπή μας και ντροπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μπλε κάρτα εκ μέρου του κυρίου Σόσνιερτ τη δέχεστε. Όχι. Δεν έχω καθόλου να συζητήσω με μισογυναίδες και ρατσιστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από αυτόν τον κύριο αρνούμε, δεν θέλω τίποτα. Δικαστικό εκ μέρους του κύριου Σόσνιες. Θα ήθελα α, να πω ότι Πρόσφατα η κυρία Γουόρτ στήριξε κάποιες κυρώσεις βάρος μου και τις υπερψήφισε. Είναι παραδεκτό να χαρακτηρίζει κάποιος ε, έτσι έναν ευρωβουλευτή και τελείως ε, αδικαιολόγητα και ε, αστήρικτα να χαρακτηρίζει κάποιον ρατσιστή και μισογίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία του Catch the Eye, μόνο ο κύριος Σουίτσα ε, θέλει να λάβει το λόγο. Ε, η κυρία, με συγχωρείτε, κυρία Σουίτσα, θέλει να λάβει το λόγο. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, ήρθε επιτέλους η ώρα να δεχτούμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το κοσυφοπαίδιο. Λυπάμαι που κάποιοι χαρακτήρισαν επαρχία το κοσυφοπαίδιο. Το κοσυφοπαίδιο είναι μια αναγνωρισμένη χώρα. Και λυπάμαι που για αμυγός εθνικούς λόγους ε, απορρίπτουν την ιδέα της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου. Νομίζω ότι ε, και η Κωσοβάρικη κυβέρνηση και οι Κωσοβάροι έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια. Έχουν ε, κυρώσει τη συμφωνία οριοθέτηση σύνορα με το Βαβροβούνιο, έχουν εντείνει τι προσπάθειε για την πάταξη διαφθορά εγκρίνοντα το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και λυπάμαι που ε, χρησιμοποιούμε αυτή τη συζήτηση για να ασκήσουμε ε, πιέσεις προς το Συμβούλιο για να επιτρέψει επιτέλους την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη νέα χώρα με τον νέο πληθυσμό. Θέλουν επιτέλους και οι, οι κατοικοί του Κωσυφοπεδίου να ταξιδεύουν ελεύθερα όπως και οι κάτοικοι των υπόλοιπων Δυτικών Βαλκανίων. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει αυτή, αυτό το αίτημα για την απαλλαγή των θεωρήσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση είναι υπέρ τη απελευθέρωση. Θα πρέπει να ασκήσουμε επίση και στο Συμβούλιο για να άρει τι επιφυλάξει του και να εγκρίνει το καθεστώ απαλλαγή. Λοιπόν, ε, τώρα ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο για να απαντήσει ο Επίτροπος κύριος Αβραμόπουλος. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν Ευχαριστώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι ευτυχής που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της επίτευξης προόδου στο φάκελο αυτό. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν πρόκειται μόνο για ε, θέμα δικαιοσύνης προς το κοσυφοπαίδιο, τις αρχές και τους πολίτες ε, αναγνώριση των προσπαθειών. Πρόκειται για σταθερότητα, πρόκειται για την ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το ευρύτερο πλαίσιο, τη μεγαλύτερη εικόνα που διακυβεύεται εδώ, ούτε την ευρωπαϊκή προοπτική όλης της περιφέρειας αυτής. Αν τους φέρομαι όλους πιο κοντά μας, θα διασφαλίσουμε και καλύτερη συνεργασία. Δεν μπορούμε ε, να ε, πιέζομαι ε, υπερβολικά κοντά στο τέρμα. Αλλιώς ρισκάρουμε το κοσυφοπαίδιο και ακόμα πιο σημαντικό οι φιλοευρωπαίοι πολίτες του να μας γυρίσουν την πλάτη και να κινηθούν προς την αντίθετη από εμάς κατεύθυνση. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν κατέστη δυνατή μία συμφωνία ε, εντός αυτής της θητείας. Ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί κατά την επόμενη το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε Επίτροπε και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Φαγιόν. Παρακαλώ Τάνια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη των σκιωδών εισηγητών και άλλων συναδέλφων που πιστεύουν ότι αξίζει στο Κωσοπαίδιο να του δώσουμε την ε, ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κοσοπέδιο δεν είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει κανείς το, τη χώρα αυτή ως κράτος αρκεί να αναγνωρίσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα ε, και η απελευθέρωση ε, ε, είναι πολύ σημαντική για τους νέους αλλά πράγματι η όλο και μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση του Κοσφοπεδίου ε, και στην απογοήτευση που θα νιώσουν οι άνθρωποι αυτοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοσοπέδιο έχει καλύψει όλε τι προποθέσει που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αναγνωρίσει το Κωσοπαίδιο, το Κοινοβούλιο επίσης και σήμερα όταν λέει κανείς ότι το Κωσοπαίδιο δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, απλά ε, ψεύδεται κανείς και συμπεριφέρεται ανεύθυνα. Καλό λοιπόν τις κυβερνήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσουν την απελευθέρωση με ειδική πλειοψηφία γιατί στο Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ομοφωνία να σταματήσει αυτό το παιχνίδι και να δράσουμε τώρα. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε για να διασφαλίσουμε την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι η τελική ψηφοφορία, είναι όμως μια σημαντική ψηφοφορία για να ε, πούμε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ξέρετε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι. Εμείς τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Εναπόκειται τώρα σε εσά να αποδείξετε την αξιοπιστία σας, να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε για τους νέους, για νέες οικογένειες, για μια νεόκοπη χώρα η οποία είναι πολύ απομονωμένη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. l'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole Manca, stato di previsione delle entrate e delle spese. Ο κύριο Μάνκα θα μιλήσει για το επόμενο θέμα, ε, για τον κατάλογο δαπανών και εσόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020. Οι υπηρεσίε μου μου λένε ότι, οι συνεργάτε μου μάλλον, μου λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι παρόν ο κύριο Μάνκα. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στο έλξ τον κύριο Ρούμπι για τρία λεπτά. Παρακαλώ, κύριο Ρούμπι. Εντάξει, προηγείται ο κύριος Μάνκα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Τι να κάνουμε. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα λαμβάνει χώρα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του Brexit. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες 48 ώρες, αλλά θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός μας πρέπει πάση θυσία να είναι έτοιμος για σκληρό Brexit, για πιο μαλακό Brexit ε, και βεβαίως και για την παραμονή των Βρετανών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που είναι βέβαια η πρώτη μας προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, αποκινούμε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάναμε διαπραγματεύσεις, πετύχαμε περικοπές, συνολικά πετύχαμε περικοπή 18 εκατομμυρίων. Ε, επιτύχαμε μία συμφωνία με το Γενικό Γραμματέα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα στην ε, επικείμενη προεκλογική εκστρατεία να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ψευδή ε, διαρροή ειδήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκε μια νέα ομάδα που μπορεί να δραστηριοποιηθεί γιατί θέλουμε γεγονότα, στοιχεία, τεκμηρίωσή τους και θέλουμε και ε, δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτά να αποτελούν τη βάση για μια ειλικρινή και διαφανή παρουσίαση των προϊόντων. Υπάρχει το εξής. Το καταστατικό των βουλευτών πρέπει και αυτό να γίνεται σεβαστό. Έχουμε το εθελοντικό συνταξιοδοτικό ταμείο των βουλευτών. Η ε, νομοθεσία υπάρχει, οι θεσμοί έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να παραμείνει αυτό το ταμείο. Εγώ δεν συμφωνώ με την απόφαση του Προεδρείου σχετικά με το τι πρέπει να γίνει με αυτό το ταμείο, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το καταποκοπή ποσό για τα έξοδα γραφείου να παραμείνει ως καταποκοπή ποσό για τους βουλευτές. Γιατί για τους βουλευτές είναι σημαντικό να μην πνιγούν μέσα στη γραφειοκρατία. Ε, βλέπουμε ότι το ε, θέμα με, τις, με τα καταποκοπή ποσά είναι ακριβώς αυτό, ότι μπορούν να βοηθήσουν στο να μην υπάρχει τόσο μεγάλη γραφειοκρατία. Αυτό που έχει σημασία είναι βεβαίως ο ίδιος ο βουλευτής να μην επιδεικνύει ανευθυνότητα στις δαπάνες. Βεβαίως πιστεύω ότι αν τελικά το Brexit πάρει μια ε, σκληρή ε, μορφή, το 6,1 των βουλευτών θα αποχωρήσει και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Ε, αυτό που με απασχολεί επίση είναι η διαφορά αμοιβών ε, στα δύο φύλλα. Οι γυναίκες βοηθοί και οι ε, υπάλληλοι πληρώνονται διαφορετικά. Όλοι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο αποτελεσματικά πρέπει να έχουν τον ίδιο μισθό. Εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο και ε, η ιατρική υπηρεσία να παίξει ρόλο στο θέμα της παρενόχλησης. Οι ασκούμενοι και αυτοί ε, πρέπει να αποζημιώνονται σωστά. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται μέσα από το επίδομα για γραμματιακά έξοδα. Τέλος, οι αντιπροσωπείες πολλές φορές είναι πολυμελείς. Οι ίδιοι βουλευτές θα πρέπει να αποφασίζουν ποιους θα παίρνουν μαζί τους σε επίπεδο βοητών, διερμηνέων. Μόνο έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε δαπάνες, γιατί πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ακόμα ε, περιθώριο να περικόψει δαπάνες. Πολύ ωραία. Τώρα για έξι λεπτά να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μάνκα. ďakujem vám pani predsedníčka za flexibilitu a za ústretovosť. vážené kolegyne kolegovia ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την κατάρτιση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο βασικό μας ρόλο, στη βασική μας αποστολή και να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους για να βελτιώσουμε το νομοθετικό μας έργο που δεν ε, συνδέεται άμεσα με την αποστολή μας θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να αποκλείεται από τον προπολογισμό. Πριν από 10 χρόνια ήμουν ο γενικός συζητητής για τον προπολογισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ίδιο ρόλο έχω και τώρα. Τότε τα κονδύλια για τη μετάφραση δεν είχαν ε, εκταμιευθεί πλήρως ε, λόγω έλλειψης προγραμματισμού και επικοινωνία και πολύ συχνά είχαμε εξωτερική ανάθεση της μετάφρασης χωρίς να έχουμε βεβαιωθεί ότι είχαμε εξαντλήσει πρώτα τους δικούς μας πόρους και ικανότητες. Μόνο για τη μετάφραση ε, εξοικονομήσαμε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έκτοτε η κατάσταση έχει βελτιωθεί ιδιαίτερω, ειδικά σε αυτό το θέμα. Αλλά και πάλι θα πρέπει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυ την διοργανική συνεργασία και το ε, δυναμικό, οι ικανότητε που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διατίθενται στη διάθεση των άλλων θεσμικών οργάνων. Έτσι θα κάνουμε οικονομίε. Γιατί δίνουμε κοινή μάχη για περισσότερη απασχόληση, ανάπτυξη και καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Μερικέ φορέ όμω μόνοι μα ε, ε, βάζουμε εμπόδια. Η ε, κοινοβουλευτική μας βοηθή ε, μερικές φορές ε, αντί να επικεντρώνονται στο βασικό τους έργο φέρονταν κατά των ευρωβουλευτών και μετά γινόταν η αξιολόγηση της δραστηριότητα κάποιων βουλευτών. 1.700 ερωτήσεις, προφορικές ερωτήσεις το χρόνο μερικές φορές είχαμε κάποιους βουλευτές να υποβάλουν με τεράστιο κόστος, γύρω στα 13 ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την επεξεργασία όλων αυτών των γραπτών και προφορικών ερωτήσεων. Ε, επίσης, δεν θα πρέπει να ε, ε, μας εκπλήσει ο χαρακτηρισμός κάποιων ερωτήσεων ως περιττών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικές φορές, παρόλο που ήταν αγαθές οι προθέσεις, το αποτέλεσμα δεν ήταν και πολύ υπεύθυνο. 9.000 ερωτήσεις προφορικές το χρόνο απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 7 εκατομμύρια θα εξοικονομούσαμε κάθε χρόνο αν το αποφεύγαμε ή αν περιορίζαμε μάλλον τον αριθμό των ερωτήσεων. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής των Προϋπολογισμών που μεγάλη πλειοψηφία ε, υποστήριξαν την ε, Δευτέρα την πρότασή μου να τεθεί ένα τέρμα στη διαδικασία των προφορικών αιτιολογήσεων ψήφου. Θα κάναμε 2 εκατομμύρια ε, ευρώ οικονομία το χρόνο και δεν θα υπήρχε λόγος να γίνεται διερμηνία για τις αιτιολογήσεις που στοχεύουν στο ε, χώρο εκλογικό σώμα. Νομίζω ότι έτσι θα μειώσουμε και το διοικητικό κόστος. Θέλουμε να μειώσουμε και τις, ε, τα ταξιδιωτικά έξοδα των υπαλλήλων ε, στις μετακινήσεις μεταξύ των τριών εδρών, χρησιμοποιώντας περισσότερο τις ε, βίντεο διασκέψεις. Επίσης, ε, θέλουμε να βοηθήσουμε τους διαπιστευμένους βοηθούς που για δύο συναπτές κοινοβουλευτικές θητείε απασχολούνται και τους λείπουν λίγες εβδομάδες ή μέρες για να τεκμηριώσουν τα δικαιώματά τους. Επίσης, θα πρέπει να καλύπτουμε και τους ασκούμενους κατά τη διάρκεια της μαθητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω και σε άλλα θεσμικά όργανα, υπάρχουν ίσω φαινόμενα ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχληση. κάτι που είναι τραυματικό, είτε είναι ε, σωματική παρενόχληση είτε ψυχολογική ηθική. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη διευκόλυνση αυτή με την παροχή ε, βοήθειας ψυχολογικής. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Επίση απλουστεύσαμε τη διαδικασία έγκριση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και σχεδόν υλοποίησαμε το στόχο μα. Ελπίζω λοιπόν ότι το επόμενο κοινοβούλιο θα συνεχίσει το έργο μας ε, και την εξοικονόμηση των κονδυλίων. Επίσης, ε, οι προβλέψεις αυτές έγιναν με βάση μια έφτακτη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν δεν υλοποιηθεί κάτι τέτοιο ή χωρί συμφωνία ή παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχε προσαρμογές στην επόμενη δημοσιονομική χρήση. Ε, η χωρίς συμφωνια η παραμεινει το ηνωμενο βασιλειο θα πρεπει να γινουν αντιστοιχε προσαρμογες στην επομενη δημοσιονομικη χρηση η ε, Βρετανοί πολίτες ε, εξαιτία παραπληροφόρησης ή ανακριβούς πληροφόρηση έλαβαν την απόφαση για την αποχώρηση. Θα πρέπει, έπρεπε να είχαν εξηγηθεί τα επιτέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θετικέ πτυχέ και οι επιτυχίες της. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει πιο κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό ξεκινήσαμε εκδηλώσει και ε, εκθέσει που θα με, περιοδικές εκθέσεις ε, στις χώρες μέλη που θα τονίζουν τα απτά επιτεύγματα της Ένωσης. Με τις κινητές αυτές εκθέσεις ε, θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και των μαθητών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ τους συνεργάτες, βοηθούς και συμβούλους μου. Εν ώψη των ευρωεκλογών ε, είχαμε ελάχιστο χρόνο, χρειάστηκε να εργαζόμαστε μέχρι αργά τη νύχτα και Σαββατοκύριακα και είχα την ανεκτήμητη συνεισφορά των βοηθών μου που άοκνα και νυχθημερών ασχολήθηκα με το θέμα αυτό παρόλο που μερικοί ξέρουν ότι δεν θα επιστρέψουν μετά τις ευρωεκλογές τους. Ευχαριστώ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και θα βρουν το δρόμο τους στη ζωή. Ε, είναι τελευταία μου αυτή η έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τελευταία μου ομιλία στην Ολομέλεια. Πάντω ήταν μεγάλη μου τιμή η συμμετοχή μου στι εργασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συνεργασία μου μαζί σα για τη δημιουργία μια καλύτερη Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε και σα ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια. Τώρα για δύο λεπτά το λόγο η κυρία gracias, Ρουβιάλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, το κύριε Μάνκα και συγχαρητήρια για το έργο σας γιατί καταφέραμε εμπρόθεσμα να ε, συζητήσουμε τις προβλέψεις εξόδων-εξόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τα 15 χρόνια και που θέτευσε ευρωβουλευτή. Και στα πλαίσια της, των επικείμενων εκλογών μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό των έργων. Τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε μια πολύ συνετή διαχείριση, κάναμε οικονομίες και προσαρμοστήκαμε στις νέες ανάγκες. Από την ανάγκη ενίσχυση της ασφάλειας των κτίριων μας, στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, των ψευδών ειδήσεων και της έγκρισης ε, ε, τη προσαρμογή, μάλλον σε μια νέα πραγματικότητα με μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 χώρε μέλη. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, μιλάμε για τον προπολογισμό τη διοίκηση ε, με αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να επιτελέσουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο. Γιατί ένα κοινοβούλιο ε, που εγκρίνει νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να έχει συμμαζέψει και τα του οίκου της. Ε, το 2013 ξεκινήσαμε μια εκστρατεία ε, με την νεολαία ζητώντας ε, για τους υποτρόφους μια αξιοπρεπή επιδότηση και χρειάστηκε πέντε χρόνια για να το καταφέρουμε. Επίσης μιλήσαμε για τη διαθέτηση του θέματος παρενόχλησης. Χρειάστηκε αρκετό χρόνος, αλλά χάρη στο κίνημα MeToo και χάρη στην δέσμευση και στράτευση πολλών ευρωβουλευτών ανδρών και γυναικών καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα κατάλογο μέτρων για να καταπολεμήσουμε την ανισότητα των φύλων. Και όταν μιλάμε για ισότητα, δεν μπορούμε στην, στο κοινοβούλιο αυτό να πρέπει να διαλέγουμε μεταξύ το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας ή μητρότητας. Γι' αυτό ζητούμε από το Προεδρείο να εφαρμόσει άμεσα ένα σύστημα που θα επιτρέπει την εξαποστάσεως ψηφοφορία, την τηλεματική ψηφοφορία, γιατί έχουμε μπει στον 21ο αιώνα, υπάρχουν οι τεχνολογίες για κάτι τέτοιο. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κούσμιουκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνοντας το λόγο στην έκθεση αυτή για την κατάσταση προβλέψεων εσόδων-εξόδων για το 2020 εκ μέρους του ECR, θα ήθελα να πω ότι θα είναι η τελευταία χρονιά του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ω εκ τούτου οι αποφάσεις και οι υποχρεώσει ε, θα πρέπει να διέπονται από την ανάγκη τη δημοσιονομική πειθαρχία και ε, το 4,34% λαμβάνοντα υπόψη ε, και την τιμαριθμική προσαρμογή του 2,5% σε σχέση με το 2019 έχουμε καταλήξει σε ποσά που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και πολύ πιστικέ οι προτάσει για τη διεύρυνση ε, της, των διπλωματικών αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Αιθιοπία, Ιδονησία και αλλού, που δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα γραφεία. Και χαίρομαι που η Επιτροπή Προπολογισμού τάχθηκε υπέρ μια και έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι, θα εξοικονομήσουμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω, αν έχουμε μόνο και μία και μόνη έδρα. Επίσης, θα πρέπει να σεβαστούμε τα κοινωνικά και συνταξιδοτικά δικαιώματα των διαπιστευμένων βοηθών, εξασφαλίζοντα του πρόσβαση σε συνταξιδοτικό σύστημα μετά από ε, δύο θητείες. Άλλωστε, και το ελεκτικό συνέδριο μίλησε για το σύστημα επικουρικής σύνταξης των ε, βουλευτών. Και μάλιστα ε, σχετικά απόφαση έλαβε και το Προεδρείο πρόσφατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει η κυρία Γιατερμάκη. Κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο ε, έχει βασικό ρόλο στον προϋπολογισμό ε, έλεγχο εσόδων και δαπανών. Ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου όμως είναι πολύ υψηλός, αν και έχουμε κάποιες εξοικονομήσεις. Η ομάδα μου ε, θέλει πάρα πολύ να υπάρχει διαφάνεια και σόφρον και χρηστή δαπάνη. Ένας τρόπος να, προάγουμε, να προαγάγουμε τη διαφάνεια είναι η κτηριακή πολιτική του Κοινοβουλίου να μην χρησιμοποιείται για γάλματα και μνημεία. Πολλές φορές ε, γράφονται ε, τα κονδύλια σε άλλη γραμμή του προπολογισμού και μετά πηγαίνουν στα κτίρια. Η κτηριακή πολιτική θα πρέπει να είναι ανοιχτή και να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Και κάτι άλλο. Ε, αυξανόμενες δαπάνες ε, για το προσωπικό τους υπαλλήλους. 6% έχουμε προαγωγές και ε, πληθωριστικές διορθώσεις. Υπάρχουν όμως και νέες θέσεις. Θα πρέπει να αποφασίσουμε πάνω σε αυτά με ανοιχτό πνεύμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον συγητή, τον κύριο Μάνκα. Ήταν ε, εύκολη συνεργασία μαζί του, όπως και με τους άλλους σκιώδεις συγητές. Και εγώ ήθελα να πω ότι ίσως είναι η τελευταία φορά που αγορεύω στο Κοινοβούλιο, διότι δεν θα υποβάλω εκ νέου υποψηφιότητα. Θα ήθελα τέλος να πω ότι οι εξοικονομήσεις και η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικά. Αν δεν τα κατοχυρώσουμε αυτά, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, μελλοντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ. Και σας ευχόμεθα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Και τώρα για 1,5 λεπτό στην κυρία Τρούπελ. Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, συνεχίζω αυτά που είπε ο κύριος Γιατεμέκη. Για μας η διαφάνεια και η ε, ετοιμότητα ε, δράσης είναι σημαντικά για τον προϋπολογισμό. Θέλουμε ένα προϋπολογισμό βέβαια για να, που θα εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα και τις καλές εργασίες του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες ε, πιστώσεις, τους πόρους. Μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο ε, αρκεί στο 2% ε, τα περισσότερα χρήματα θέλουμε να τα δίδουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες για καλά προγράμματα και όχι προς ίδιον όφελος. Πολύ σωστή σκέψη. Όμως πρέπει όλοι να μπορούμε να εργαζόμεθα αποτελεσματικά και τονίζω θα πρέπει να υπάρχει εσωτερική ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των ομάδων, ημών των βουλευτών, αλλά και της διοίκησης. Δηλαδή αν υπάρχουν υπερβολικές εντάσεις στο σύστημα δημιουργούνται ε, προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Επίσης, με όλες τις φιλοδοξίες που μπορεί να διατυπώσει το Κοινοβούλιο σε σχέση με τα απαιτούμενα κονδύλια, για παράδειγμα στις μεταφραστικές υπηρεσίες ε, όταν δεν χρειαζόμαστε κάποιες γλώσσες δεν χρειάζεται να τι δηλώνουμε και εξοικονομούμε χρήματα έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τα ταξίδια. Ε, ε για εύλογους λόγους ε, θέλουμε να επικεντρώνουμε τις αντιπροσωπείες σε συγκεκριμένα ταξίδια. Ε, επίσης, ε, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε εισιτήρια business όταν είναι μικρές οι αποστάσεις. Ε, αυτό είναι σημαντικό και στο τέλος ε, θα μας εξασφαλίσει και τα κονδύλια που χρειαζόμαστε για να εργαζόμεθα σωστά. Ο κύριος Βέγγας δεν είναι εδώ. Προχωρώ τον κύριο Βάλλη για δύο λεπτά. Ε? Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι η δημοκρατία πολύ σωστά έχει και δαπάνε το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το κόστος της δημοκρατίας, αλλά η διασπάθηση που λαμβάνει η χώρα στη δημοκρατία. Και σε αυτό το κοινοβούλιο ε, αυτά τα πέντε χρόνια διαπιστώσαμε διασπάθηση χρημάτων από κονδύλια, τα οποία δίδονται για διεύρυνση, αλλά και για ε, κόμματα, για πολιτικά κόμματα. Μιλάμε για 63 εκατομμύρια ευρώ 360 συνολικά περίπου εκατομμύρια, τα οποία δόθηκαν στα πολιτικά κόμματα. Σε γενικές λοιπόν γραμμές, ε, ο προπολογισμό περνάει το 1 δις 700 εκατομμύρια, περίπου στα 2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς ε, να κάνει μια σωστή πολιτική εκστρατεία, να λέει στους πολίτες ότι πρέπει να κάνουμε οικονομίες αλλά ε, επειδή θα υπάρξει και το Brexit θα υπάρχουν και λιγότεροι ευρωβουλευτές. Αυτό το κοινοβούλιο παρόλα αυτά συνεχίζει τις δαπάνες και τις πατάλες. Ε, με τέτοια κατάσταση δυστυχώς ο δεν υπάρχει μέλλον για αυτό το κοινοβούλιο. Ο κύριος ε, Έλισεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για τις δαπάνες και τα έσοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνολικά το Κοινοβούλιο έχει 2 δισεκατομμύρια για τον προϋπολογισμό του και έχει και 4 εκατομμύρια έξτρα, ε, δηλαδή προστίθενται και άλλα εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα είναι απαραίτητα έτσι ώστε να ε, συνεχίζει η κατακυδεμόνευση του Ευρωπαίου πολίτη, να δημιουργείται υποτίθεται η ευρωπαϊκή συνείδηση. Ε, Υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά κέντρα και κινητές εγκαταστάσεις ε, στα κράτη-μέλη, ακριβά γραφεία και η προπαγάνδα που λαμβάνει η χώρα και αυτή είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά εκείνο για το οποίο δεν μιλάμε είναι για την μεγάλη απειλή στις ευρωπαϊκές αξίες. Γιατί μην ξεχνάτε κυρία Πρόεδρε, πολλοί τυχοδιώκτες έρχονται σε εμά με ολέτριες συνέπειες. Το μυσαλόδοξο Ισλάμ δεν μπορεί να συμβαστεί με τις δικές μας ευρωπαϊκές αξίες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον εξισλαμισμό, είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Πάω τώρα πίσω στο σχέδιο του προϋπολογισμού γίνεται λόγος για το ότι χάσαμε μία ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να περικόψουμε τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Δεν, ε, γιατί δεν μειώνονται οι μισθοί των υπαλλήλων, γιατί δεν μειώνεται αυτά, μειώνονται αυτά τα καταποκοπή ποσά και σε τελική ανάλυση τι θα γίνει και με αυτή την συνταξιωτική ρύθμιση για τους βουλευτές. Και αυτό κοστίζει πάρα πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φροντίζει πολύ καλά τον εαυτό του, ε, προσλαμβάνει συνεργάτες ε, οι οποίοι παραδείγματο χάρη αποσπώνται στην ε, Ασία, στη Δυτική Αφρική. Είναι απόλυτη παράνοια κυρία Πρόεδρε. Επίκυνται οι εκλογές και έχει έρθει πλέον η χρονική στιγμή έτσι ώστε να τιμωρηθεί αυτή η ελίτε που υπάρχει στην Ευρώπη έχει έρθει η στιγμή να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή. Ευχαριστώ κύριε Φερνάνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή ε, αποχαιρετώντα τον, να τον ευχαριστήσω για την πολύ στενή συνεργασία και το πολύ καλό μα έργο. Σίγουρα ποτέ δεν είναι εύκολο να καταρτίζει κανεί έναν προπολογισμό, πολλό δε μάλλον ιδιαίτερα σε μία προεκλογική περίοδο. Γι' αυτό είναι διπλάσια τα συγχαρητήρια προς τον ε, Βλαντιβίρ Μάνκα και σε όλους τους ε, σκιώδεις που συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης. Το ΕΛΚ ήταν ανέκαθεν υπέρ της ε, διαφάνειας και της Χρηστή διαχείριση. με τα απαραίτητα όμω ε, μέσα και πόρους για να τα στο κοινοβουλευτικό μας έργο. Γιατί μερικές φορές ε, μια κακή νομοθεσία έχει τεράστιο κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και κάναμε μεγάλη προσπάθεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια προσπάθεια που προϋποθέτει την ποιότητα των υπηρεσιών και επαγγελματίες υπαλλήλους. Έχουμε πραγματικά πολύ ποιοτικέ υπηρεσίες και εξαιρετικούς υπαλλήλου και ο στόχος να μειώσουμε στο μέγιστο, στο έπακρο τις δαπάνες δεν θα πρέπει να ε, γίνει βάρος των αρχών που έχουμε, όπως είναι η αρχή της πολυγλωσσίας. Θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να εκφράζεται στη γλώσσα του, στη μητρική του γλώσσα. Χρειαζόμαστε και μετάφραση, χρειαζόμαστε και διερμηνία. Σίγουρα μπορούν να γίνουν κάποιες οικονομίες, όπως έγιναν στον τομέα αυτό, αλλά όχι εις βάρος της ε, αρχής της πολυγλωσσίας. Επίσης είναι προφανές ότι έχουμε ε, το Παρλαμεντάριο, έχουμε τον Νίκο της Ευρώπης, έχουμε γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε κράτος μέλος. Όλα αυτά έχουν κόστος. Αλλά έτσι όμως μπορούμε να προβάλλουμε το έργο μας και να προβάλλουμε την ευρωπαϊκή ιστορία και τις αξίες μας και τις αρχές μας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της χρηστής διαχείρισης της ε, δημοσιονομικής πειθαρχία, της διαφάνειας και των ε, ελάχιστων αλλά απαραίτητων και επαρκών μέσων για να τα απεξέλθουμε στο κοινοβουλευτικό μας έργο και να το επιτελέσουμε με αριστεία. Ευχαριστώ δύο λεπτά κύριος Χάουαρθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Βλάντιμιρ Μάνκε για το έργο του ως, εισηγητής, ως εισηγητή. Και επειδή είναι εξαιρετικός συνάδελφος και τα τελευταία δύο χρόνια στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ήταν πολύτιμος ε, ε, συνάδελφος. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 31 που αναφέρεται στο θέμα της ε, κοινοβουλευτικής των βοηθών, των διαπιστευμένων βοηθών. Ε, πολλές φορές, ε, επειδή η εκλογική θητεία είναι λίγο μικρότερη, δεν φτάνουν στα 10 χρόνια για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ελπίζω να κατοχυρωθεί αυτό. Επίσης, ε, οι εκπαιδευόμενοι στα δεν πρέπει να εργάζονται ε, δωρεάν, αμυστοί, ε, και βέβαια όλοι θα πρέπει να εργάζονται χωρίς παρενοχλήσεις ε, σεξουαλικές και άλλες. Ε, το κοινοβούλιο μας λέγουν είναι δαπανηρό, αλλά συγκρίνεται πολύ θετικά σε σχέση με το, τη Βουλή των Αντιπροσώπων ε, για παράδειγμα στην Ευρωπα... στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημοκρατία έχει το τίμημά της και αν ε, αυτό το τίμημα δεν είναι ούτε 4 ευρώ αναπολίτη αναχρόνο, ε, τότε έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη γι' αυτό. Βεβαίω και μπορούμε να κάνουμε πρόοδους, να καταργήσουμε τη δεύτερη έδρα. Θα μπορούσαμε να ε, προχωρήσουμε με τη βοήθεια των βουλευτών. Και πιστεύω ότι πολύ σημαντικό είναι το πολύ γλωσσικό κοινοβούλιο να συνεχιστεί και θα πρέπει να μπορούν ε, οι βουλευτές μας να απευθύνονται στους πολίτες της Ένωσης. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να καταργήσουμε την ε, μετάφραση. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, διότι όταν εξετάζομαι μόνο τα δημοσιονομικά και όχι την σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Μισελ Ντεπρέ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρά την ποιότητα του έργου του κύριου Μάνκα, του εισηγητή μας που θέλω να συγχαρώ και τον, να συγχαρώ και τον σκηνοδόν εισηγητών, δεν σας κρύβω ότι είμαι βερδεμένος για τη συμφωνία αυτή που επετεύχθη με την Επιτροπή Προπολογισμών. Φυσικά και σημειώνω τη μείωση 18 εκατομμύρια ευρώ που πέτυχε η Επιτροπή Προπολογισμών σε σχέση με την αρχική πρόταση του Γενικού Γραμματέα που ενέκρινε το Προεδρείο. Προσωπικά πιστεύω ότι η μείωση αυτή δεν φτάνει. Το ποσοστό αύξηση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε, δεδομένων των νέων αναγκών και έκτακτων αναγκών, να είναι στο επίπεδο του πληθωρισμού. Και όταν βλέπω ότι οι επιστώσει για τι αμοιβέ του προσωπικού αυξάνουν κατά 6% του χρόνου, αναρωτιέμαι είτε στην ποιότητα των προβλέψεων που γίνονται σε σχέση με τον πληθωρισμό δηλαδή, είτε αναρωτιέμαι τι μας κρύβεται σε αυτή την αύξηση. Και υπάρχουν και δύο άλλα πράγματα που με απασχολούν. Πρώτα απ' όλα, η πρόθεση του Κοινοβουλίου να αυξήσει τι δραστηριότητέ του και τι διπλωματικέ του σχέσει με διάφορε χώρε, για παράδειγμα στην Ινδονησία και την Αιθιοπία. Και ενώ υπάρχουν πρεσβείες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτέ τι χώρε. Και υπάρχει και την προσώπευση που κοστίζει και πολλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξωτερική δράση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κερδίσουμε αν ενισχύσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου εκεί. Και αντίθετα με τον συνάδελφο Μάνκα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πολλαπλασιάζουμε και τα κέντρα ε, που δημιουργούνται σε διάφορες χώρες που είναι κάτι σαν κάτι μίνι παρλαμεντάριου που θέλουμε να οργανώσουμε και να εγκαταστήσουμε σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αναγκαίο και το καταλαβαίνω να έχουμε αποτελεσματικού μηχανισμού για να ενημερώνεται ο πολίτη για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τι προτεραιότητε που υποστηρίζει αυτό. Όμω προτιμάω να επενδύσω στου ανθρώπου και όχι στου τείχου στον πετών. Στου δημοσιογράφου, για παράδειγμα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι ο πολλαπλασιασμός των ε, τούβλων. Ο κύριος Στάραντ, ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπω συμβαίνει συνήθω στην Επιτροπή Προπολογισμών, πάντα συμφωνώ με τον κύριο Τεπρέ, οπότε και τώρα με αυτά που τον άκουσα να λέει. Όμω, επιτρέψτε μου να προσθέσω ένα σημείο. Ευχαριστώντα βέβαια τον κύριο Μάνκα για τη στήριξή του, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να έχουμε τόσα θέματα μπροστά μας. Οπότε μπράβο κύριε Μάκη, ευχαριστώ. Περισσότερη δουλειά για τις πολιτικές ομάδες. Αυτό ακριβώς είναι που γίνεται και έγινε όταν ήμουνα και εγώ εισηγητής. Θέλουμε 36 παραπάνω θέσεις για τις πολιτικές ομάδες και έχοντας καλά καμουφλάρει τα πράγματα τελικά τα κατάφεραν. Όμως ακριβώς αυτό είναι το οποίο οδηγεί σε διάφορα Brexit, η κίτρινα γυλαίκα κλπ. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι ας αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και ας περιορίσουμε τις ορέξεις των διαχειριστών των κομμάτων. Αλλιώς δεν θα φτάσουμε στα, στις υψηλές προδιαγραφές της ελεύθερης εντολής των ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά ο κύριος Άρνοτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή ε, θα λέγατε ότι δεν είναι δικιά μου δουλειά αφού έρχεται το Brexit, αλλά ε, και όμω, διότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συνεισφέρει στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει παράγραφο 25, η οποία μιλάει για το σταμάτημα αυτού του τσίρκου που ταξιδεύουμε κάθε μήνα στο Στρασβούργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμω σε διάφορε εκθέσει ψηφίζει από διάφορε επιτροπέ κάθε χρόνο, τη μία μετά την άλλη, ξανά και ξανά και ξανά παρόλα αυτά καμία αλλαγή δεν γίνεται. Είμαστε εδώ γιατί τελικά ποιος αποφασίζει, όχι και αυτή είναι η διαφορά. Με την Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα στη συζήτηση. Η έκθεση αυτή λοιπόν